Good afternoon to everybody. Back again all... Καλησπέρα σας. Καλώς επιστρέψατε μετά την τυρκουάζη εβδομάδα και ελπίζω να μην έχει και κανείς προβλήματα με τον ιό. Να ξεκινήσουμε αυτή αμέσως με την ημερήσια διάταξη. Πρώτον, έγκριση αυτής, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι είναι εγκεκριμένη ως έχει επί τα ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω μερικέ. Πρώτα απ' όλα, οι αποφάσει των συντονιστών τη 18η Φεβρουαρίου βρίσκονται στους φακέλους σα για τη σημερινή συνεδρίαση και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει. θα θεωρηθούν εγκεκριμένε. Δεύτερο σημείο. Μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του κορονοϊού, του περίφημου COVID-19. Όπω τα γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο έχει λάβει κάποια μέτρα πρόληψη σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19. Τα μέτρα αυτά αφορούν τα μέλη και του υπαλλήλου του Κοινοβουλίου, καθώ και επισκέπτε υποσκεκλημένου που έρχονται στι εγκαταστάσει του σώματο. Να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα μέτρα που εγκρίθηκαν και ότι θα ακολουθήσετε τι συστάσει που έχουν δοθεί. και πάλι σε σχέση με τον κορονοϊό, τρίτη εισαγωγική παρατήρηση για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 24 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο βοήθεια ε, για να στηρίξει τα κράτη-μέλη και τι διεθνεί προσπάθειε ώστε να επιβραδυνθεί η εξέπλωση του ιού. Το πακέτο έχει αξία 232 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατομμύρια θα τα πάρουμε από την ενεργοποίηση του Ταμείου Επίκουσας Βοήθειας. Μεταφορ... Αιτήματα μεταφορών θα υποβληθούν κατά πάσα πιθανότητα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το πακέτο αποτελείται από τα εξής τέσσερα ε, σημεία. 114 εκατομμύρια για να υποστηριχθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ιδίω η ετοιμότητα και η απόκριση ε, διεθνώς με ένα διεθνές πρόγραμμα. Τα 15 εκατομμύρια ε, προβλέπονται για την Αφρική για να υποστηριχθούν μέτρα όπως η ταχεία διάγνωση και η επιδημιολογική η επιδημιολογική ε, παραεπιφυλακή. 100 εκατομμύρια είναι το τρίτο στοιχείο της βοήθειας αυτής, κατεπηγόντως απαραίτητα για την διάγνωση, την θεραπεία και την πρόληψη. 90 εκατομμύρια εκ των 100 θα προέλθουν από την εταιρική σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες και τελευταίο στοιχείο, 3 εκατομμύρια για τον επαναπατρισμό και τις πτήσεις Ευρωπαίων πολιτών από την Γουχάν ε, μέσω του ε, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Πολιτικής πολιτικής προστασίας. Θα έχετε λάβει την επιστολή του Επιτρόπου Χάν με όλες τις λεπτομέρειες που αναλύουν το ζήτημα αυτό. Και τέταρτο σημείο μεταξύ των ανακοινώσεων, τελευταία ανακοίνωση για σήμερα από πλευρά. μου. Παρακαλώ. Μπορούμε να έχουμε την επιστολή. Ναι, θα αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές, αν δεν έχει ήδη αποσταλεί. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ης Φεβρουαρίου. Κύριε Άντρες. Ναι, με συγχωρείτε, έχω αναγνώσει την επιστολή, αλλά έχω κάποιες απορίες για κάποια σημεία της επιστολής. Πρώτα απ' όλα, για το τμήμα που αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για αυτό που αφορά την ε, συνεργασία με τις φαρμακοβιομηχανίες την ε, εταιρική σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Θα μπορούσαμε να έχουμε περαιτέρω πληροφορίε για αυτό από την Επιτροπή πώς μπορούμε να οργανωθούμε. Ε, όχι αναγκαστικά ευθύ αμέσω, έστω και γραπτέ απαντήσει. Απλώ θα ήθελα περισσότερε λεπτομέρειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται εδώ, βλέπω να γνέφηκα τα φατικά. Παρακαλώ, αν θέλετε, απαντήστε. Ναι, μπορούμε να αποστείλουμε γραπτές απαντήσεις στην ερώτηση που τέθηκε. Θα ενημερώσω σχετικά τη γραμματεία σας. Κύριε Άντερσεν, Ε, θα μπορούσε ο κύριος Άντερσεν να σα αποστείλει τι ερωτήσεις του μέσω της γραμματείας για να λάβει και τις απαντήσεις. Ωραία. κάποιο άλλος. Συνεχίζω λοιπόν με το τέταρτο σημείο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 20 Φεβρουαρίου. Το δελτίο ενημέρωσης για τα δημοσιονομικά, για τον προπολογισμό, συμπεριλαμβάνει τις απόψεις των ε, ε, μελών της Δημοκρατικής Ομάδας του Κοινοβουλίου για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια ε, τελική έκβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Υπήρχε δογματική στάση εκ μέρους κάποιων ηγετών, κάποιοι, ακολούθησαν μια στάση στενόμυαλη λογιστών αντί να συζητήσουν σημαντικά στρατηγικά σημεία πολιτικής. Και ε, παγιδεύτηκαν σε εθνικιστικές ε, απόψεις με προτεραιότητες δικές τους εσωτερικές προτεραιότητες στην πρόταση που είχαμε επιτάπητος μαζί με το non-paper που είχε υποβάλει ως πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν λάβαμε καμία θετική άποψη και καμία έγκριση. Ήταν ε, ασυνεπής η στάση των ηγετών και θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι απλώς να έχουμε περισσότερες περικοπές από τη μία και λιγότερες προτεραιότητες από την άλλη. Δεν είναι αυτό που θέλουμε ως επιτυχημένη λύση. Γι' αυτό μια τέτοια προσέγγιση δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τις μετατροπές που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προπολογισμού απαραίτητα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για τις προκλήσεις συγχρηματοδότησης και τις διεθνείς προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν θα υποστηρίξει αυτή τη στάση το Κοινοβούλιο. Έχω προσκαλέσει τον Επίτροπο Χάν στην επόμενη συνεδρίαση Επιτροπή στι 19 Μαρτίου για να συζητήσουμε του λόγου που φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο και βεβαίω να δούμε τι ε, εξέλιξη θα μπορούσε να έχει όλη την πραγμάτευση. Μετά την αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η έναρξη των νέων προγραμμάτων ε, είναι έτσι κι αλλιώ de facto αργοπορημένη και εάν βρεθεί συμφωνία τον Μάιο ή τον Ιούνιο, πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί αν είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μπορούμε παρόλα αυτά να επιτρέψουμε πάυση των προγραμμάτων τρέκου στι 31 Δεκεμβρίου και γι' αυτό απευθύνουμε διαρκώ έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα άμεση ανταπόκριση ε, στην ε, έκτακτη αυτή ανάγκη για να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώ αρνείται και επανειλημμένω έχει αρνηθεί ε, να, συνεχίσει να ασκεί πιέσει για να βρεθεί συμφωνία. Τώρα όμω μα τελειώνει ο χρόνο που έχουμε στη διαθέσή και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνθηκών κάτι να κάνει και να υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο εναλλακτική λύση ω ε, πρώτη κίνηση. Και το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μόλι την περασμένη εβδομάδα και με το πόσο έκτακτε ανάγκε έχουν παρουσιαστεί, θα το ξέρετε ότι ήταν δύσκολη η εβδομάδα ω προ τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Άκουσα ότι ο έχει μειώσει δραστικά τι ε, θετικέ εκτιμήσει για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Και σε αυτή τη χρονική συγκυρία να σερνόμαστε τώρα με ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ αρνητικό. Γιατί όχι μόνο πλήττει την ε, εμπιστοσύνη που θέλουμε να έχουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοιες οικονομικές, χρηματο, ε, συνθήκες, αλλά γιατί επί της ουσίας θα έπρεπε να στηρίξουμε και να συμβάλλουμε στην στήριξη τη οικονομία μα. Η περασμένη εβδομάδα πραγματικά μα δίνει επιπλέον επιχειρήματα για να συνεχίσουμε να εντείνουμε την πίεση και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Και αν όχι, να είμαστε έτοιμοι για ένα εναλλακτικό σενάριο, για ένα εναλλακτικό σχέδιο με κατεπήγοντα μέτρα, εφόσον δεν υπάρξει τελική συμφωνία. Είναι ε, άκρο επιτακτική ανάγκη. Θέλει κανείς να σχολιάσει από αυτού. The silence Η σιωπή σας προς απάντησή μου φαντάζομαι ότι σημαίνει συμφωνία. Ωραία. Να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Δημοσιονομικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σημείο 3. Το σχέδιο έκθεση είχε υποβληθεί και συζητηθεί στη συνάντησή μα στι 22 Ιανουαρίου. Και προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, να σα πω ότι η τροπολογία 157-157 έχει αποσυρθεί. Να κάνουμε πρώτα απ' όλα μια δοκιμή για τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε, παρακαλώ. Ψηφίσατε άπαντες πέρας. Μου λένε ότι υπάρχει ένας περάριθμος στους σοσιαλιστές. Συνεχίζει να υπάρχει ένας παραπάνω στους σοσιαλιστές ή φταίει το μηχάνημα. It's okay. It's okay. Εντάξει τώρα. Εψήφισαν άπαντε πέρας. Πρώτα απ' όλα. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Συγγνώμη. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, για την 51 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, λήξη. Απορρίπτεται. 16 κατά, 12 υπέρ. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική πτά, Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 19 προς 11. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84 Β. Υπέρ. 84 β υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. 84 β. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125. Υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε την 125. Λοιπόν, τροπολογία 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστή 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξει. Απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. συμβιβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 210 Β. Περ. Κατά. Αποχές. Γκρίνετ. 212. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνετ. Συμβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνετ. Τροπολογία 2.14. Περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.16. Υπέρ. Κατά. πρέπει να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 221 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38. 39 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 1, στο εκτιμώντας EB, 1 α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εικόν 1β, υπέρ, συγγνώμη, καταπίπτει. Εικόν 2α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκόν, 13 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έκον 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στο ψήφισμα, στην ψηφοφορία όλης της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε άρχεται ψηφοφορία ονομαστική λήξει. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στον κύριο Κορμό. Thank you. Σας ευχαριστώ. There are uh, under points 4, 5 and... Σημεία 4, 5 και 6 σχετικά με τις μεταφορές στο τμήμα 3 και στα άλλα τμήματα και όσον αφορά την πολιτική κτηρίων δεν έχουμε κάτι. Επομένως ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας. Then on the building policy. Σημείο 7. Για την ε, κτηριακή πολιτική επίσης δεν έχουμε λάβει κάποιες πληροφορίες. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως που αφορά εκτιμήσεις ε, εσόδων και δαπανών για το δημοσιονομικό έτος 2021, τμήμα 1 και θα δώσω αμέσως ε, τον λόγο στον εισηγητή κύριο Ολιβιέ Σαστέλ, έτσι ώστε να μας παρουσιάσει το προσχέδιο έκθεση σχετικά με τα θέματα αυτά για το έτος 2021. Κύριε Σαστέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο έκθεσης το οποίο σας παρουσιάζω σήμερα εγγράφεται ε, σε δύο, στη σειρά δύο ακροάσεων που είχε ε, ναι, γίνει με τον ε, υπεύθυνο του αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου ήδη το Φεβρουάριο του 2020. Ξέρετε ότι ακόμα βρισκόμαστε στο προηγούμενο πι ε, ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει γιατί δεν έχουν ορκηθεί οι ε, για την περίοδο 2021-2027 και δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς ε, τα στοιχεία για την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως θα πρέπει να ξαναδούμε τι θα γίνει με την πλήρη και σωστή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κινητικότητα, κτίρια, αμοιβέ κλπ. Γνωρίζουμε ότι για το σε 2021 προβλέπονται 2 δις 120 εκατομμύρια ε, ευρώ. Έχουμε 72 ε, εκατομμύρια αύξησης, εκ των οποίων 32 αφορούν ε, συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις. Θα ήθελα επίσης ε, να επιστήσω την προσοχή σας και στο εξής. Οι προβλέψεις για τα έτη 18, 19 και 20 αντιπροσώπευαν αντιστοίχως αύξηση 2 και 30, 2 και 48 και 2,68% κάθε φορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πράγμα που σημαίνει ότι οι προβλέψεις όσον αφορά τις ε, δαπάνες που υποβάλλεται ε, από τον Γενικό Γραμματέα ε, είναι οπωσδήποτε σε σωστά πλαίσια. Πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε συνεκτικοί, αξιόπιστοι, προσεκτικοί να ε, ε, ακολουθούμε τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης και οπωσδήποτε να προωθούμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί στις ακροάσεις. Επομένως είναι σημαντικό να αναλυθούν δεόντως οι διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού και οι περικοπές του προϋπολογισμού ε, που θα μας επιτρέψουν ωστόσο να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τον τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ επίσης ε, και στις ε, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit, μια και υπάρχει περικοπή του προϋπολογισμού λόγω έλλειψης των εισφορών της χώρας αυτής. Είναι γεγονός ότι ήδη στο 2020 είχε εγγραφεί αυτή η μειωτική τάση και εκπλήσωμε που το 2021 δεν αναφέρεται ας πούμε η γραμμή για τις ε, μετακινήσεις ε, των βουλευτών δεν ε, έχει μειωθεί από το 18 στο 21. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ξαναδούμε γιατί δεν προκύπτει η εξοικονόμηση μετά από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να ξαναδούμε. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα είναι το πρασίνισμα του Κοινοβουλίου καθώς επίσης και οι, βιώσιμες, οι βιώσιμοι στόχοι και πρέπει να είναι σαφές ότι όταν ας πούμε το Κοινοβούλιο ε, θέτει κάποιους ε, ενεργειακούς ε, στόχους εξοικονόμησης ενέργειας όπως είναι η μείωση της χρήσης του χαρτιού και λοιπά, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να προσπαθεί να τις υλοποιήσει. Επίσης πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να διευρύνει την πολιτική στάθμευση στο κεντρικό κτίριο που ισχύει δηλαδή στο κεντρικό κτίριο στο σύνολο ε, των κτίριων του Κοινοβουλίου, κυρίως ε, να ε, προωθήσει την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, ε, θα μπορούσε να ε, προωθήσει περισσότερο τρόπους όπως ε, η τηλεδιάσκεψη, video conference και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μειώσει τα αεροπορικά εισιτήρια. Επίσης γνωρίζουμε ότι θα πρέπει, πρέπει να περιοριστεί αυτή η μετακίνηση κυβωτίων από την μία έδρα του Κοινοβουλίου στην άλλη. Φυσικά θα πρέπει να ξαναδούμε την επικοινωνία εκεί μας πολιτική πρέπει οπωσδήποτε να στραφούμε προς τους ε, νέους. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα ε, για το διετές, ε, τη διετή εκδήλωση για τους νέους της Ευρώπης που θα προβλέπει το έτος πριν αλλά και το έτος μετά μια σειρά ανταλλαγών και επισκέψεων με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ε, δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να στεγαστούν οι νέοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Επίσης ε, η κτηριακή πολιτική είναι πολύ σημαντική. Ε, συζητήσαμε και θα ξανασυζητήσουμε οπωσδήποτε αυτό το θέμα του mopping up transfer το οποίο αφορά την κτηριακή πολιτική και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφασίσουμε να το χρηματοδοτήσουμε και πώς θα χρηματοδοτήσουμε και τις σχετικές επενδύσεις. Επίσης, ε, το κτίριο Πόλο Αρισπάκ ε, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, αναμένονται αποφάσεις, έτσι ώστε να ληφθούν κάποιες διατάξεις όσον αφορά ε, την αξιολόγηση, καθώς επίσης και τη σωστή κατανομή αναθέσει των των ε, διαφόρων κονδυλίων. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τεχνικές λύσεις έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι βουλευτές να μπορούν να ψηφίζουν όταν έχουν άδεια μητρότητας, ε, γονική ή ε, υγείας. Επίσης, στην γνωμοδότησή μου θα αναφερθώ και στον εκφοβισμό και την παρενόχληση ηθική ή άλλου είδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό ε, να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αξιολόγηση των νέων διαδικασιών που έχει θέσει σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δούμε πώς οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν ακόμα καλύτερα να προσαρμοστούν ε, στην ζωή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα τελειώνοντας να αναφερθώ σε δύο άλλα θέματα. Πρώτον, το θέμα της επικοινωνίας αλλά και της πληροφορικής όσον αφορά την επικοινωνία. Το είδαμε και στις ακροάσεις. Ακούστηκαν πολλές νέες ιδέες ε, με στόχο το Κοινοβούλιο να επικοινωνεί καλύτερα και περισσότερο. Ε, ας πούμε το κέντρο Europa Experience ξέρουμε ότι ε, και για το 20 και για το 2021 όλες ε, οι πρωτεύουσε μέχρι το 2024 θα έχουν τη διαδικασία αυτή. Είναι καλό για το Κοινοβούλιο. Επίσης πρέπει να γίνει η αξιολόγηση αντικτύπου όσον αφορά τις δαπάνες και την ταξινόμηση και των δαπανών συγκεκριμένα και για το 2021. Ε, επίσης ε, ε, να δούμε αν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν κάποιες κινητές δομές στο Παρλαμεντάριο. Και εδώ έχουμε πολλές δυνατότητες και εναλλακτικέ ως Κοινοβούλιο έτσι ώστε και καλά να γίνουν και χωρίς να είναι πολύ δαπανηρά. Επίσης η διπλωματική εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου εκτός της ενώσεως εγώ θα ήθελα ε, να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία ε, της εκπροσώπησης ε, του Κοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε, δύο, σε τρία άλλα μέρη, έτσι όπως έχει προβλεφθεί από απόφαση του Προεδρείου. Για να τελειώσω, θα αναφερθώ στην πληροφορική. Είναι γεγονός ότι η ασφάλεια πρέπει και να, να είναι και να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα. Εκπλήσω γιατί οι γραμμές αυτές ε, οι πέντε δηλαδή γραμμές πληροφορικής ε, βλέπουν μια αύξηση 20 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις. Μας ε, εξηγήθηκε σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρξει υβριδικός εξοπλισμός που θα αντικαταστήσει ε, κάποια παλαιότερα στοιχεία και θα υπάρξει εξοικονόμηση αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ελπίζουμε όλοι. Πάντως με αυτή η ιδέα ε, της ε, ανάπτυξης ενός εργαλείου που θα είναι σε θέση να μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο όλες τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι πριν ξεκινήσουμε μια τέτοια περιπέτεια θα πρέπει να έχουμε πραγματικά σωστή ανάλυση αυτού του ενδεχομένου και αυτού αυτού του θέματος. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως παραμένω στην διάθεσή σας. Ε, ελπίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες που θα ολοκληρώσουμε την έκθεση θα πρόκειται για μια έκθεση ισορροπημένη ε, και μέχρι τις 11 Μαρτίου στη μία το μεσημέρι θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι ενδεχόμενες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ίνσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την έκθεση. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε, όμως πραγματικά λυπούμε που δεν πήραμε όλες τις απαντήσεις που θέλαμε στις ερωτήσεις μας ως τώρα. Προετοιμάζουμε ήδη τροπολογίες για την ερχόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές και πλούσιες συζητήσεις. Mr. Thank you κύριος Κόζακοφ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ενημέρωση θεωρώ ότι έχουμε κάποια ζητήματα και πολιτικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα για τον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά για το Κοινοβούλιο. Ω προ την πολιτική διάσταση, δεν ξέρω αν από οποιαδήποτε προοπτική μπορούμε να επιτρέψουμε το Κοινοβούλιο να χρηματοδοτείται περισσότερο από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Έχουμε Brexit, έχουμε ε, την ανάγκη να πείσουμε του πολίτε μα ότι πρέπει να παραμείνουν ε, ε, πιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα να αυξήσουμε σε ασυνήθιστα επίπεδα τον προπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου και για το 2021 από δημοσιονομική σκοπιά πρέπει να αναφέρω ότι ακόμα δεν έχουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε αν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα τα προγράμματά μα ή όχι ε, για το μέλλον. Α πούμε για την κτηριακή πολιτική. Θα έλεγα ότι το, για το Polar Risk Pack υπάρχουν. Ε, κάποια σχέδια, αλλά θα ήθελα να δω πολύ περισσότερα, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια που προγραμματίζονται για το χρόνο, για το κτίριο αυτό, για την προοπτική τη πενταετία που θέλουμε να έχουμε, να δούμε και άλλε προτάσει πριν κάνουμε την επιλογή. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερη κατανόηση για το τι θα γίνει ε, με τα κτίρια και από την σκοπιά του προπολογισμού που να λάβουμε υπόψη ότι πολλές φορές αυτά που δεν έχουν ταπανηθεί στο τέλος της χρονιάς με το ραμασάζ ε, χρησιμοποιούνται για τα κτίρια, αξιοποιούνται δηλαδή τα προηγούμενα έτη, αλλά και εκεί χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Και για το ραμασάζ το είδαμε ε, για την ε, μεγαλύτερη ε, χρηματοδότηση που θέλουμε να έχουμε για τα, για τα προγράμματα συντήρησης και για το αν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα κέντρα για τα παρλαμεντάριου στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε με το 2024. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν πώ θα φέρουμε πιο κοντά το βορρά στο νότο και την Ανατολή στη Δύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθουν πιο κοντά μα οι πολίτε. Για την ε, τεχνητή ευφυα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα gadget, μ' αρέσει και η τεχνολογία, αλλά δεν ξέρω αν τα επόμενα 5-6 χρόνια θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ε, προηγμένες μεταφραστικές λύσεις, όχι από τα αγγλικά στα γαλλικά, αλλά από τα λιθουανικά στα κροατικά, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό και δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα να επενδύσουμε τόσο πολύ σε αυτά, χωρίς να είμαστε από την αρχή σίγουροι ότι κάτι θα μας προσφέρουν εξελίξεις αυτές τις τεχνολογίες. Και πάλι όμως θα σας ευχαριστούμε για το σχέδιο της έκθεσης και που συμπεριλάβατε πολλά από τα θέματα που απασχολούσαν τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποιος από τους ID Ähm, Η εκπρόσωπο τη ID δεν βρίσκεται εδώ, γι' αυτό θέλω να μιλήσω εγώ στη θέση τη. Για την έκθεση αυτή που και εγώ την βρίσκω πολύ καλή και ευχαριστώ γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση που δεν μιλάμε για τον προπολογισμό για το ε, ΣΠΑ και μιλάμε για το 3,5% που θα αυξηθεί και ότι έχουμε και ε, μια αύξηση 2% που δεν φαίνεται να έχει ε, θεμελιωθεί σε σοβαρά επιχειρήματα. Δεν φαίνεται πολύ λογικό αυτό για τον προπολογισμό. Ιδίω επειδή υπάρχει το γεγονό ότι έχουμε πλέον λιγότερα μέλη στο Κοινοβούλιο. Αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστούμε. Κάποιο από τους Πρασίνους. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, κύριε Γιόνσα. E, e, e, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο εισηγητή. Βέβαια έχουμε κάποιους άγνωστους παράγοντες και δεν ξέρουμε τι άλλο θα εμφανιστεί σύντομα σε σχέση με το τι θα γίνει το 2021. Ο προπολογισμό του πρέπει να είναι στοχευμένος σε πραγματικά προβλήματα, ρεαλιστικός και αποτελεσματικός. Και νομίζω ότι όλοι αναμένουμε να έχουμε καλή διαχείριση καλή διοίκηση και υποστηρίξη στο προσωπικό μας. Δεν θέλουμε λοιπόν περικοπές στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γνωρίζει προς τα που θα στραφεί, πώς θα, ποια πορεία θα ακολουθήσει, γιατί ακόμη και οι ούροι άνεμοι δεν θα μας βοηθήσουν. Θα πρέπει να ξέρει λοιπόν προς τα που θα βάλει πλώρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Κάποιο άλλο μέλος θέλει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν ε, να πάρω το λόγο το θέμα αυτό, το συζήτησα με τους συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που νομίζω ότι είναι ουσιαστικά και τα έχω απογραμμίσει και σε προηγούμενε συζητήσει. Καταρχήν, ε, το θέμα τη επικοινωνία, που υπογράμμισε και ο Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μα ε, και φυσικά βελτιώνοντας ε, τις ε, παροχή πληροφοριών σε σχέση με το τι κάνουμε στις ε, εθνικές εκλογές μας περιφέρειες. Αλλά θα πρέπει να απευθυνθούμε και στην Ευρωπαϊκή Διασπορά. Έχουμε όλο ένα και περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται από μία χώρα στην άλλη, ψηφίζουν στις ευρωεκλογέ στη χώρα κατοικίας, αλλά και στην πατρίδα τους. Στις τελευταίες ευρωεκλογέ λόγου χάρη, εκατομμύρια Ευρωπαίοι ψήφισαν στην Ρουμανία, στη χώρα μου έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια ομάνους που ψήφισαν ε, ε, υποψήφιου από τη Ρουμανία, ακόμη και αν ζουν ε, σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, να έχουμε πόρους για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και για τα γραφεία του Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη, για να ενημερώνουν για αυτή τη νέα κατηγορία θα πρέπει να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί σε ευρωεκλογέ. Του αρέσει η Ευρώπη, υποστηρίζουν ε, την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε για τα νέα εργαλεία επικοινωνία. Και ένα δεύτερο θέμα που θα πρέπει να υπογραμμιστεί περισσότερο είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στι ε, δαπάνε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ αναφέρουμε στις συμβάσεις, στους προμηθευτέ και πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αν είμαστε διαφανείς θα έχουν οι πολίτες περισσότερη εμπιστοσύνη σε εμά. Και φυσικά, καθώ μιλάμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε όλη τη συζήτηση για τον επόμενο προπολογισμό, θα πρέπει εμεί να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Γιατί αν τα καταφέρουμε, τότε ίσω ε, μπορούμε να πείσουμε και τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σαστέλ, για το σημαντικό έργο που έχει υλοποιήσει και να υποστηρίξω τις ανησυχίες του σε σχέση ε, με την παρουσίαση αυτού του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην δώσουμε το την εντύπωση ότι ο προπολογισμό είναι για μα, αλλά ότι είναι για του πολίτε. Ε, σε σχέση με το θέμα τώρα τη έκθεση, ε, για το θέμα των κτηρίων. Θέλω επίσης ε, να χαιρετήσω τα διάφορα στοιχεία ανάλυσης που περιλαμβάνονται στο κείμενο μεταξύ των σημείων 18 και 25 της έκθεσης. Θέλω να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι το σημείο 19, το θέμα της συντήρησης των κτηρίων, προκειμένου να είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ, γιατί βάζουμε στην ίδια γραμμή του προπολογισμού διάφορα έργα διαφορετικής φύσης. Και αν το επιτρέπει συνάδελφος Σουζεκόφ, θέλω να υπογραμμίσω και εγώ πόσο σημαντικός είναι ο πολιετής προγραμματισμός για τις εργασίες, για τα έργα, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο. Και αν συμφωνείτε, Πρόεδρε, ίσω κάποια στιγμή θα μπορούσε να παρουσιαστεί αυτό στην Επιτροπή Προπολογισμού, γιατί σήμερα ε, ουσιαστικά παρακολουθούμε μεμονωμένα τα διάφορα έργα. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη παρουσίαση σε ό,τι αφορά και το κτίριο ΣΠΑΚ. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες γιατί ε, δεν υπάρχει υποχρεωτική πληροφόρηση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Τον ευχαριστώ για την εξαιρετική του εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία του και για το μέλλον και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο σε αυτή την έκθεση θα μπορέσει να συμφωνήσει πάνω σε κεντρικά σημεία, σε σημεία κλειδιά. Γιατί συζητούμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Συμφωνούμε με το ένα σημείο φέτος, μετά την επόμενη χρονιά κάνουμε μια διαφορετική συμβιβαστική λύση. Και Υπάρχουν όμως ένα σωρό πράγματα που θα πρέπει να τα δούμε μία και καλή, γιατί οι πολίτες δεν γνωρίζουν όλη αυτή την διοίκηση και το κόστος ε, και δεν ξέρουν ότι όλο αυτό αφορά λιγότερο από 7% του συνολικού προϋπολογισμού. Νομίζουν ότι είναι πολύ περισσότερο τμήμα του προϋπολογισμού. Ε, το θέμα είναι τι πρέπει να έχουμε. Το ελάχιστο που ε, είναι ικανό και αρκετό. Γιατί καλό είναι να κάνουμε ε, έτσι ε, δημο ε, μικροπολιτική ας το πούμε, αλλά να σας πω ότι ήταν ας πούμε πάρα πολύ δύσκολο να βάλουμε Wi-Fi, ίντερνετ στο Στρασβούργο και αν τώρα ας πούμε λέγαμε θα κόψουμε το Wi-Fi, τι θα γινότανε ή ας πούμε ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας με μεγάλη δυσκολία προχώρησε. Ε, τώρα όλοι λένε «Α, θετικό είναι αυτό». Ε, το θέμα της ε, διερμηνίας, της μετάφρασης, αυτό κοστίζει. Αλλά χρειαζόμαστε ανθρώπους, χρειαζόμαστε προσωπικό που να είναι ποιότητος, που να είναι αξιόλογο και αξιόπιστο. Επομένως, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε να μην θεωρήσουν οι πολίτες ότι όλο αυτό είναι υπερβολικά ακριβό για τους πολίτες. Εμείς εδώ νομοθετούμε. Ο στόχος ε, είναι ε, να υπάρχει μία νομοθετική ε, αριστεία. Είναι ένας στόχος τον οποίο θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι. Και μετά έρχονται βεβαίως τα κτίρια και τα λοιπά, τα οποία φυσικά και αυτά κοστίζουν χρήματα. Όσον αφορά τώρα τις παραδοσιακές ας πούμε ερωτήσεις για τους λαϊκιστές ε, και που πολλές φορές τις συζητούμε ακόμα περισσότερο και στον ε, προϋπολογισμό τμήμα 3 ε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία, να επιτύχουμε μία συμφωνία έτσι ώστε να υπάρξει ε, συμβιβασμός μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων, τουλάχιστον των φιλοευρωπαϊκών μονάδων και να γίνει μία συζήτηση, μία και καλή και να μην αλλάξει οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι, όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαστέλ ε, για να, κάνει, να εξάγει τα τελικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε Τάχιστα, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσει και τα σχόλιά του και τις προτάσεις τους. Προφανώς θα φροντίσω να λάβω υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσει. και Πολύ σύντομα, νομίζω μεθαύριο, έχουμε μια συνεδρίαση όλων των συντονιστών, των ε, σκιωδών, ε, για να συζητήσουμε τα θέματα της έκθεσης, αλλά για να δούμε και το ποσό των χρηματοδοτήσεων, τις ενδεχόμενες περικοπές, επειδή η πρότησή μας θα πρέπει μετά να ε, περάσει από τη συμφωνία του Προεδρείου. Θα έχει τη μορφή συνεδρίασης συνδιαλλαγής 19 και 20 Μαρτίου τρέχοντος. Και προτού ε, περάσουμε σε έκθεση τεχνικής τροπολογίας που ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί στις 30 Μαρτίου και από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Προτού περάσουμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια 1η Απριλίου στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να ε, ολοκληρώσω λέγοντας ότι ανάλογα ε, σε σχέση με τις διάφορες παρεμβάσεις που άκουσα κατανοώ ότι συνολικά είναι ε, σημαντικό να υπάρχει αύξηση και να δούμε βεβαίως τι γίνεται συγκριτικά και με τα προηγούμενα χρόνια. Ε, πέρσι, για τον προπολογισμό του 2020, η συνδιαλλαγή όρισε την αύξηση σε 2,68% νομίζω ήταν 18,5 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την εκτίμηση που είχε κάνει ο Γενικό Γραμματέα πρόπερση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώ από την ίδια αρχή. Δηλαδή να δούμε όλε τι δημοσιονομικέ γραμμέ για να φροντίσουμε να είμαστε και δραστικοί και αποτελεσματικοί και συνεπεί και να υπάρχει δουλειά. Ε, γιατί αν θέλουμε να μπορούμε να κοιτάξουμε τη δουλειά μας ε, τώρα μελλοντικά, το, να κοιτάξουμε λοιπόν τον προπολογισμό που θα μας αποτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτόν που θα αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, δείχνοντας μια πολύ σοβαρή στάση στον δικό μας τον ίδιο τον προπολογισμό. Να σας θυμίσω ότι οι τροπολογίες σας ε, αναμένονται μέχρι τις 11 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αστέλ είπε ήδη ε, ποιε είναι οι σημαντικέ ε, ημερομηνίε, τα ραντεβού μα, για να είμαστε βέβαιοι όμω ότι όλοι κατάλαβα, να τι ξαναπώ. Ε, υποβολή τροπολογιών 11 Μαρτίου, έκθεση στην Μπάτ 30 Μαρτίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στο, στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Τελευταίο σημείο για την ημερήσια διαταξή σήμερα, σημείο 9, η συμφωνία σύμπραξη στον τομέα τη βιώσιμη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας των Σέιχελών. Κύριε Χριστοφόρου, έχετε το λόγο. Ε, η σημερινή συμφωνία... Η σημερινή συμφωνία που συζητάμε είναι σύμπραξη στον τομέα τη βιώσιμη αλληλεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία των Σιχελών. Υφίσταται από το 2007. Απλά τώρα συζητάμε την προέκταση του εξαετούς πρωτοκόλλου, το οποίο έληξε τον Ιανουάριο και ουσιαστικά συζητάμε την εφαρμογή νέου πρωτοκόλλου και συμφωνίας από το 2020 μέχρι το 2026. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής της δράσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, της γνωστών ACP, για να δημιουργήσει αυτήν την στήριξη όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των αλλιευτικών αποθεμάτων σε αυτήν την περιοχή. Λαμβάνοντα ταυτόχρονα όμω, και είναι πολύ σημαντικό, υπόψη και τι δημοκρατικέ αρχέ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η νέα συμφωνία δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα. Στόχο, είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δημοκρατία ε, των Σεχελών για στενότερη συνεργασία στη βιώσιμη αλληλεία με σκοπό την πρόθεση μιας υπεύθυνη εκμετάλλευση αλληλευτικών πόρων. Δεύτερο, να υπάρξει μια καλύτερη και προώθηση όσον αφορά πιο αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία στον τομέα τη αλληλεία. Επίση, λήφθηκαν υπόψη και να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και αξιολογήσει ε, των ειδικών οι οποίοι ορίστηκαν και ήταν ανεξάρτητοι ειδικοί εμπειρογνώμονε ε, επί του θέματο. Η υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτά τα πλαίσια τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ω αντιπαροχή προ αυτή τη συμφωνία είναι η παραχώρηση ποσού ύψου 5.300.000 ευρώ ετησίω. Οφείλω να επισημάνω και τελειώνω τα δύο πολύ σημαντικά. Ότι πρώτον, η νέα συμφωνία ορίζει τη σύσταση μειχτή επιτροπή η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου 2026 και δεύτερον, η Επιτροπή Προπολογισμού καλεί την αρμόδια και καθήλυν Επιτροπή Αλληλεία, όπω προωθήσει προψήφιση το Ευρωκοινοβούλιο και εγκρίνει το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία ω Σιχελό. Thank you Thank you. Mr. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σε επίπεδο προπολογισμού δεν έχω πολλά να πω, όμως η Επιτροπή Αλίας ε, θα πρέπει να ε, ελέγξει το πώς ε, θα δοθούν αυτά τα κονδύλια και το πώς θα δαπανηθούν. Γιατί είχαμε ε, κάποιες ειδήσει ε, στη Γαλλία που μας ε, είπαν ότι αυτά τα κονδύλια ε, κυρίως ε, πήγαιναν ε, για την κατασκευή ενός λιμανιού που χρησιμεύει για τον ελληνισμό των ευρωπαϊκών πλοίων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτός ο έλεγχος και να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες του τοπικού κλάδου. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι δαπανώνται αυτά τα κονδύλια όπως πρέπει. Αυτή είναι μια ανησυχία που έχω εγώ και θέλω να την αναφέρω. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε διαδικασία συγκατάθεσης, δεν υπάρχουν τροπολογίες και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 18 Μαρτίου. Και αυτή είναι η ημερομηνία και της επόμενης συνεδριασής μας 18 και 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και 30 του μήνα στο Στρασβούργο σε έκτακτη συνεδρίαση. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρίασή μας στο Επανειδή.